Κυρίες και κύριοι, ας αρχίσουμε αν συμφωνείτε τις εργασίες μας και σας παρακαλώ κάνετε ησυχία. Όποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να συζητούν μπορούν να το πράξουν εκτός εθούσης. Αρχίζει λοιπόν η διακοινοβουλευτική συνάντηση, η διακοινοβουλευτική διάσκεψη και ευχαριστώ τον πρόεδρο Βαν Ρόμποη καθώς και τον πρόεδρο Βαρόσο, τον Αντιπρόεδρο κύριο Πιτέλα του Κοινοβουλίου που ε, θα υποδεχθεί τα πρόσωπα αυτά εκ μέρου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και τους συναδέλφους Ευρωβουλευτές που δέχθηκαν την πρόσκλησή μας να έλθουν να συμμετάσχουν στην διακοινοβουλευτική αυτή διάσκεψη που αποτελεί και μια πρώτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβρη αποφάσισε να προτείνει την συμπλήρωση της νέας διαδικασίας που απεικλήθη ευρωπαϊκό εξάμεινο με την εισαγωγή των, της δυνατότητας συναντήσεων μεταξύ όλων των εκπροσώπων των Εθνικών Βουλών, όλων των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών που έχουν σχέση με οικονομικά, με δημοσιονομικά και με κοινωνικά θέματα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή της κυρίας Μπάουλς, η, της κυρίας Μπερέζ και η δική μου των προϋπολογισμών τις οποίες έχω την τιμή να ηγούμε, καθώς επίσης και οι αρμόδιες συναρμόδιες, μάλλον οι κοινοβουλευτικές επιτροπές των Εθνικών Βουλών, που κατά κάποιο τρόπο η σημερινή διάσκεψη αποτελεί ένα πρώτο βήμα της διαδικασίας του άρθρου 13 της νέας συμφωνίας για τα δημοσιονομικά που προβλέπει τον συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών των χωρών που συνυπογράφουν την συμφωνία αυτή. Η κρίση απέδειξε πράγματι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε δημοσιονομικές πολιτικές απομονωμένοι, ο καθένας για τον εαυτό του. Κατέδειξε επίσης η κρίση ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτική συμφωνία αποτελεσματική και βιώσιμη μόνο στις διασκέψεις κορυφής, είτε ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή της Ζώνης Ευρώ, εάν δεν υπάρχει και μια στήριξη κοινοβουλευτική και μια συζήτηση κοινοβουλευτική. Γνωρίζω ότι οι πρόεδροι Βαν Ρομπόη και Μπαρόσο έχουν επιμείνει επ' αυτού και έχουν κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε με την ολομέλεια αυτή όπου θα λάβουν το λόγο οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων. Μετά θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο κύριος Βαν Ρόμποη που θα είναι υποχρεωμένος να φύγει στις θα ακούσει τις πρώτες ερωτήσεις και στο πρώτο μισό του απογεύματος θα χωριστούμε σε δύο εργαστήρια που το ένα θα ασχοληθεί με τη δημοσιονομική πειθαρχία και το άλλο περισσότερο με την στήριξη της ανάπτυξης. Προβλέπεται και δείπνο εργασίας υπό την Προεδρία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σούλτς. Σήμερα το βράδυ λοιπόν και αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε για να δούμε πώς εκκινώντα από τη νέα συνθήκη ιδίω θα μπορέσουμε να θεμελιώσουμε, να βάλουμε σε λειτουργία αυτά τα νέα εργαλεία για να ξεκινήσουμε ξανά, να τονώσουμε και πάλι την οικονομική ανάκαμψη. Σας ευχαριστώ και πάλι και δίνω το λόγο ευθύ αμέσω στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Τζάνι Πιτέλα, που εκπροσωπεί τον πρόεδρό μας, κ. Σούλτς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Λαμαζούρ, και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσους βρίσκονται εδώ ε, στο όνομα του Προέδρου Σούλτ αλλά και προσωπικώ ε, θα ήθελα να χαιρετήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον κύριο Φαν Ρομπόη, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κύριο Μπαρόζο και Πρέπει να αιτιολογήσω την απουσία του Προέδρου Σούλτσου που είναι ε, δεσμευμένο σε άλλες συνεδριάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τελευταίες εξελίξεις ε, στην οικονομική κρίση, η σημερινή συνεδρίαση αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία. Έχουμε την ευκαιρία εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το σπουδαίο θέμα του οικονομικού συντονισμού στην Ευρώπη. Η πείρα που έχουμε μέχρι στιγμής και τα σφάλματα που έγιναν κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ετών της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ιδιαίτερα τα σφάλματα που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ε, κατέστησαν προφανή την ανάγκη για πιο αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αντιπροσωπεύει βεβαίως ε, το σωστό πλαίσιο για να... την επέτευξη αυτού του στόχου, ιδιαίτερα για τι χώρε. Ε, της Ευρωζώνης που συνδέονται με κοινέ ευθύνε. Η σημερινή συζήτηση θα χρησιμεύσει βεβαίω να εξεταστούν δύο σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Πρώτον, η ανάγκη τη εξασφάλιση τη πλήρου δημοκρατική νομιμότητα μια τέτοια διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, για να το πούμε ξεκάθαρα, να το πούμε στα ράτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν μπορούν να εξαιρούνται από οποιαδήποτε επιλογή που αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Δεύτερον, η ανάγκη να εγγυηθούμε αποτελεσματικό συντονιστό και όχι μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Συμβούλιο σε σχέση με μια συνταγή κατά της κρίσης που βασίζεται τόσο στην μείωση του ελλείμματος και πολύ λιγότερο στις πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη. Πολύ στην ακαμψία όσον αφορά την δημοσιονομική πειθαρχία και πολύ λίγο βασίζεται σε μέσα για να στηριχτούν ένα μεγάλο πλαίσιο επενδύσεων που θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναζωογονηθεί. Αγαπητέ Πρόεδρε Βανορομπόη, αγαπητέ Πρόεδρε Μπαρόζο, ε, τα, γεγονότα μας δείχνουν ότι οι περιορισμοί, οι περικοπές του προπολογισμού δείχνουν ότι περισσότερο πλήττουν τις οικονομίες στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πέρα από το να απαντήσουν στη λογική της πλήρους ε, Δημοκρατική νομιμότητα, θα έχουν έτσι την ευκαιρία να δώσουν μια αναπάντηση στην κρίση που θα είναι πιο ε, κοινώ αποδεκτή και πιο αποτελεσματική κατά τη γνώμη μου. Η πολιτική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικής πολιτικής αντιπαράθεσης και το σωστότερο βήμα για να γίνει μια τέτοια αντιπαράθεση είναι αυτό εδώ. Για να λυθεί ένα τόσο λεπτό ζήτημα, θα πρέπει βεβαίως να εξεταστούν ε, οι λογαριασμοί, αλλά και να ανεβάσουμε τους στόχους μας, να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Και γι' αυτό και θεωρώ πως θα πρέπει να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσω να εγγυηθεί ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώνονται μέσα στο πλαίσιο μεταρρύθμισης των εθνικών πολιτικών θα μεταφράζονται από κοινού σε ένα επίπεδο που θα είναι επαρκώς ε, προσαρμοσμένο ώστε να επιτευχθούν οι πρωτογενείς στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τις χώρες που δεν ε, επιτυγχάνουν τις δεσμεύσεις όσον αφορά την εναρμόνιση για την εσωτερική αγορά και να χρησιμοποιήσει δεσμευτικές μεθόδους και καταναγκαστικές μεθόδους ώστε στη διάρκεια της ε, ολοκλήρωσης των διαφόρων τομέων όπως των μεταφορών της ενέργειας να προχωρήσουμε και να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις όσον αφορά τους φραγμούς στην ενιαία αγορά. Χρειάζεται να υπάρχουν δεσμευτικοί και φρέσκια, φρέσκοι πόροι, όπως ε, τα ευρωομόλογα και ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Φαρομπόη, κύριε Μπαρόζο, ε, Πρόεδρε Λαμασούρ, θα πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομία της Ευρωζώνης και της Ένωσης εν γέννη. Η επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων που παρατηρούμε δίνουν σαφώς το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε και γρήγορα την ατζέντα μας, στοχεύοντας με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα και φιλοδοξία προς την ανάπτυξη. Και ελπίζω πως ε, μπορούμε να θεωρήσουμε την επιστολή που έχουν υπογράψει 12 επικεφαλής κυβερνήσεων και έχουν ε, παραλείπτει εσά, Πρόεδρε Φανοπόη, θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για μια νέα πορεία. Ευχαριστώ και καλή δουλειά σε όλους. Ευχαριστώ κύριε θα ήθελα να πω σε όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση ότι αν έχουν ερωτήματα να θέσουν στους προέδρους, στους ομιλητές του πάνελ, θα πρέπει να υποβάλουν γραπτά ερωτήματα. Σας έχουμε διανύμει έντυπα, κάποια τα έχετε ήδη συμπληρώσει, ούτω ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε σωστά τη συζήτηση. Και ζητώ από τον κάθε ένα από εσά να, μην να μην ξεπεράσει τα τρία λεπτά. Τον πρόεδρο... Το λόγο έχει ο πρόεδρος Φαν Ρομπόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διακεκριμένα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Το ότι έχετε συναντηθεί εδώ σήμερα και θα συναντηθείτε και αύριο είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι οι καιροί αλλάζουν και ότι οι εθνικές πολιτικές ε, συγκεράνεται όλο και περισσότερο με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η ευρωπαϊκή κοινότητα υπήρχε στο παρελθόν σε ένα πλανήτη μόνο και οι εθνικές ε, πολιτικές εφαρμόζονταν σε 6, σε 9, σε 15 ή και παραπάνω διαφορετικούς πλανήτες. Έτσι ήταν τα πράγματα στο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν τελειώσει σήμερα, διότι η κρίση με το εθνικό δημόσιο χρέος έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό είναι πρόβλημα καθημερινό, όλων μας. Και έτσι η Ευρώπη δεν είναι μια μεγάλη ιδέα αφηρημένη που θα λάβει σάρκα και οστά στο μέλλον. Είναι καθημερινή εμπειρία και καθημερινή καθημερινό βίωμα για όλους μας. Η αλληλεξάρτησή μας είναι περισσότερο σαφής παρά ποτέ. Εξού και περισσότερο σαφής παρά ποτέ είναι η συνυπευθυνότητα θεσμικών οργάνων και κυβερνήσεων για να ξεπεράσουν την κρίση, συνυπευθυνότητα και από πλευράς εθνικών κοινοβουλίων επίσης. Από την έναρξη της ε, ελληνικής κρίσης, ε, τα γεγονότα και οι εξελίξεις μας ανάγκασαν να λάβουμε ε, σοβαρές αποφάσεις και οι ηγέτες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρειάστηκε να αναλάβουν δράση από κοινού. Ενεπλάκησαν όλο και περισσότερο ε, στις καθημερινές δραστηριότητες της Ευρωζώνης. με τις συνεχείς διαπραγματεύσεις του τελευταίου πακέτου στήριξης της Ελλάδας, τα χρήματα του φορολογουμένου ήταν αυτό το οποίο αποτελούσε το διακύβευμα και γι' αυτό είχαμε τα κατάλληλα όργανα και τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο και συμμετείχε πολύ έντονα στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις για την εξάδα μέτρων, την νομοθετική δέσμη για την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κερδίζουν όλοι η... Ό,τι συμβαίνει στη Σλοβακία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, αλλού, ε, το παρατηρούμε από παντού στην Ευρώπη και μας ενδιαφέρει όλους. Τα εθνικά κοινοβούλια με ένα συγκεκριμένο τρόπο έχουν μετατραπεί σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το το φαινόμενο της πολιτικής αλληλεξάρτησης. Οι αποφάσεις ενός έχουν επιπτώσεις σε όλους. Η έλλειψη αλληλεγγύης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την Ευρώπη, όπως σε κίνδυνο τη έτη η έλλειψη δημοσιονομικής σταθερότητας. Οι πιστότριες χώρες πρέπει να συνεργαστούν με τις οφειλέτριες χώρες. Όλοι έχουμε αυτό το κοινό εγχείρημα το οποίο πρέπει να φέρουμε σε πέρας και πόσο μάλλον οι χώρες που είναι μέλη της ζώνης ε, του ευρώ για αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να υπονομεύεται το κοινό καλό. Ορισμένοι με πολύ απορριπτικό τρόπο θεωρούν ότι τα γεγονότα διαμορφώθηκαν με αυτόν τον τρόπο διότι οι ηγέτες της Ευρώπης έδρασαν για το κοινό καλό μόνο λόγω της πίεσης των γεγονότων και όχι γιατί το πίστευαν πραγματικά. Ε, και έτσι να είναι πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ καλό και ε, άντλησαν οι ηγέτες τα διδάγματα από την κρίση. Ε, όταν ε, χρειάστηκε ε, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, το έπραξαν. Καταρχάς τα χρήματα που διακυβεύονται είναι πολλά και αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η, κρίση του εθνικού χρέους όπως και η κρίση των τραπεζών το 2008 απαιτεί χρήματα του φορολογουμένου με τη μορφή δανείων και εγγύσεων. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι σχετικά μικρός, περίπου 1% του ΑΕΠ. Δεν μπορούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δράσουν από μόνα τους. Επομένως, είναι απαραίτητο να παρέμβουν οι χώρες μέλη. Μιλούμε για 500 δις ή για άνω του 5% του ΑΕΠ της, χω... ζώνης του ευρώ. Και εξού και οι αποφάσεις χρειάστηκε να ληφθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Πάρα πολλοί πρωθυπουργοί θα προτιμούσαν ε, τα θέματα αυτά να είχαν αποφασιστεί σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Οικονομίας ή Οικονομικών ωστόσο χρειάζονταν χρήματα. Αυτό κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο, σε καιρούς κρίσης φτάνουμε στα όρια των θεσμικών οργάνων τα οποία έχουν ε, οικοδομηθεί με συγκεκριμένη διάρθρωση. Έχουμε εισέλθει σε αχαρτογράφητη περιοχή και θα πρέπει ε, νέοι κανόνες να θεσπιστούν. Με 27 ηγέτες χωρών μελών, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλοι ε, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι και ο καθένας διαδραματίζει το ρόλο του. Δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι από αυτή την κατάσταση. Ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες νιώθουν παραμερισμένοι. Άλλοι είναι, λένε ότι η παραδοσιακή κοινοτική μέθοδος έχει εγκαταληφθεί. Ε, για όλα αυτά έχω να πω το εξή. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να ζήσουν μαζί με αυτή τη νέα αλληλεξάρτηση και παρόλο που έχουν αναλυθεί νέοι ε, διακυβερνητικοί ρόλοι, η δουλειά που έχει παραχθεί, το προϊόν που έχει παραχθεί, έχει οδηγήσει σε πιο ισχυρούς κεντρικούς θεσμούς. Και θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει άνευ προηγουμένου εξουσία εποπτείας. Ε, το δικαστήριο θα ελέγξει την ε, ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της δέσμης όλων αυτών των μέτρων. η ραχοκοκαλιά ε, του όλου εγχειρήματο είναι αυτή η εξάδα μέτρων που αποκαλείται six-pack. Έχει λοιπόν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση και γι' αυτό έχει συσταθεί μια task force, μια ειδική ομάδα. Έχουμε ε, το ε, plus Pact που είναι η θελούσια δέσμευση από χώρες που είναι μέλη του ευρώ και χώρες που δεν είναι μέλη. Όλα αυτά ε, θα προσκομίσουν αποτελέσματα εντός ε, του συνήθους ευρωπαϊκού πλαισίου. πλαισίου. Όσον αφορά στις δημοσιονομικές πολιτικές, όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Έχουμε εργαστεί σκληρά για να ευθυγραμμίσουμε τις νομοθεσίες αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται. Ε, Πολύ συχνά τα κράτη-μέλη καθορίζουν ένα κατόφλι μαζί ως προς το έλλειμμα και το χρέος σε επίπεδο ευρωπαϊκό και ατομικά αποφασίζουν πώς θα συλλέξουν ε, χρήματα, θα συγκεντρώσουν έσοδα και πώς θα τα δαπανίσουν. Έτσι, τα εθνικά κοινοβούλια διατηρούν την δημοσιονομική ε, εθνική κυριαρχία για όσο χρόνο οι επιδόσεις δεν απειλούν τη δημοσιονομική σταθερότητα του συνόλου της Ευρώπης. Έτσι, οι χώρες με υπερβολικό το έλλειμμα θα συνάψουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθεί το έλλειμμα ε, κάτω από το κατόφλι του 3% σε σχέση με το ΑΕΠ. Ωστόσο, ορισμένοι εθνικοί πολιτικοί νιώθουν κάπως άβολα με τα νέα καθήκοντα και εγχειρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι κάθε πλευρά της πολιτικής ζωής αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. Κάθε ε, εθνικός βουλευτής θα πρέπει να ενδιαφέρεται να συνομιλεί με συναδέλφους του ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο αλλά και ομολόγους του σε κοινοβούλια άλλων κρατών μελών. Ένας μέλος της Γερμανικής Βουλής, της Bundestag, μπορεί βεβαίως να ωφεληθεί πάρα πολύ ομιλώντας με Ιταλό συνάδελφό του, Έλληνα ή Σλοβάκο. Με τη νέα συνθήκη έχουν θεσπιστεί συσκέψεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το φόρουμ ε, που, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ όλοι και είμαστε παρόντες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην λαμβάνονται αποφάσεις, ωστόσο διαμορφώνονται απόψεις και ε, εδρεώνονται ο διάλογος. Εύχομαι να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Πολύ συχνά ως εξωτερικός παρατηρητής είχα στο παρελθόν την εντύπωση ότι σε διαφορετικούς κόσμους ζούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τα Εθνικά Κοινοβούλια ενδιαφέρονταν συνέχεια και περισσότερο για εγχώρια ζητήματα και ε, ήθελαν να πατήσουν περισσότερο φρένο ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να δώσει ορμή και να ανεβάσει το ρυθμό της ταχύτητας ως προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ε, έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, του 2012. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη φετινή χρονιά. Έχουμε τη μελέτη της Επιτροπής από τον Νοέμβριο του 2011. Με τις μεταρρυθμίσεις ε, θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία μέχρι τον Ιούνιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας κυρίως με τη θέση σε ισχύ της νομοθετικής δέσμης για την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης, της εξάδας αυτής των μέτρων δηλαδή. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά δεν ισχύουν στον ίδιο βαθμό για τις χώρες που δεν είναι ε, μέλη της ζώνης του ευρώ. Οι κυρώσεις δεν ισχύουν για τις χώρες αυτές. Η Επιτροπή παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κύκλους των κρατών μελών που ε, βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και γνωμοδοτη και έτσι εσείς στα Εθνικά Κοινοβούλια έχετε περισσότερες ευκαιρίες να κάνετε καλύτερο διάλογο με τις εθνικές κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμείνου η Επιτροπή αξιολογεί και μακροοικονομικές πολιτικές μεγαλύτερου βεληνικούς. Ε, αποφάσισε να συντάξει περισσότερες εκθέσεις για ε, χώρες που έχουν συγκεκριμένες ανισορροπίες, όπως ε, πλεονάσματα στο ισοζύγιο πληρωμών, π.χ. η Σουηδία. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις στις χώρες να διορθώσουν, να αποκαταστήσουν αυτού του είδους τις ανισορροπίες. Ή δελώς μπορεί να δοθεί λαβή για κυρώσεις. Όλος αυτός ο καινούριο τρόπος δουλειάς αντικατοπτρίζει τις καινούργιες ευρωπαϊκές εξελίξεις μετά την κρίση. Ό,τι συμβαίνει σε μία χώρα επηρεάζει τις γειτονικέ και κυρίως ε, όταν μιλούμε για τη ζώνη του ευρώ. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ε, σε θέματα δημοσιονομικά αλλά και σε θέματα εργασιακού δυναμικού θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη πριν από την υιοθέτηση οποιασδήποτε μεταρρύθμιση σε επίπεδο ε, φορολογικό, δημοσιονομικό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο η μεταρρύθμιση στη μία χώρα θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά ε, τις υπόλοιπες. Όλοι για έναν και ένας για όλους λοιπόν. Είναι ευθύνη των εθνικών ε, κοινοβουλίων να προσαρμοστούν σε αυτή την καινούργια κατάσταση. Πολύ συχνά λέγεται ότι εμείς αποφασίζουμε και κλεισμένων των θυρών. Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση ή κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν θα πάρει σημαντικές αποφάσεις ε, κάτω από τα φώτα των προβολέων της δημοσιότητας. Ωστόσο, όταν παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις, έχουμε αφοκραστεί πολύ προσεκτικά ε, τις ανάγκες όλων. Στις ε, δικές μας συσκέψει νιώθουμε την παρουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων τα οποία εσείς εκπροσωπείτε. Ακούμε ε, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έναρξη της συνεδρίασής μας, έναν πρόεδρο στον οποίο λογοδοτεί άμεσα ο πρόεδρος Μπαρόζο και πολλοί εθνικοί ηγέτες αναφέρονται στη θέση του Κοινοβουλίου της αντίστοιχης χώρας όταν ε, παίρνουν το λόγο για να υπερασπιστούν συγκεκριμένη τροπολογία επί του κειμένου. Θέλω να σας πω ότι είμαι μόνο στην αίθουσα που δεν έχω ε, κοινοβούλιο. Ε, πρώην πρόεδρος Εθνικού Κοινοβουλίου, είναι η αλήθεια ότι μου λείπει αυτό πάρα πολύ. Έχω ψηφοφόρους, αλλά είναι μόνο 27 αυτοί που με εκλέγουν. Είναι 27 ψηφοφόροι αυτοί που με εκλέγουν, οι οποίοι είναι και δημοκρατικώς εκλεγμένοι οι ίδιοι. Αγαπητά μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα 60 χρόνια ολοκλήρωσης και ενοποίησης μας έχουν δείξει ότι η Ευρώπη ε, χτίζεται μέσα από μια αργή διαδικασία η οποία συχνά ε, μπορεί να πατήσει πάνω σε βατήρα για να ε, προχωρήσει πιο γρήγορα. Έχουμε όμως φτάσει σε μεγάλο επίπεδο εμβάθυσης και σήμερα πλέον η Ευρώπη είναι μέρος των εθνικών, των εγχώριων πολιτικών. Εξού και έχει εξαιρετική σημασία να οργανώνονται διάλογοι όπως ο διάλογος που έχει οργανωθεί σε αυτή την αίθουσα εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μετά από την σημερινή συνάντηση θα αισθάνεστε λιγότερο απογοητευμένος, έχετε μπροστά σας όλη αυτή την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το λόγο θα λάβει τώρα ο, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόσο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα παρόν στην έναρξη της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και χαίρομαι για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οργανώσει την παρούσα συνάντηση και ιδιαίτερα επειδή θα έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις και με εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων που με εφαρμόζοντας τις μεταρρυθμίσεις επιτόπου παίζει βέβαια ένα ζωτικό ρόλο. Η διακοινοβουλευτική συζήτηση είναι πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική σε δράση. Πιστεύω ότι είναι ουσιώδες να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή δημοκρασία, δημοκρατία συγγνώμη, με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εθνικών δημοκρατικών διαδικασιών και της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διαδικασίας. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ένας τρόπος για να προλάβουμε τις επικίνδυνες πολιτικές ανισορροπίες πριν επεκταθούν σε άλλες χώρες και έτσι είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής μας προσέγγισης για την επίλυση της κρίσης και της προσπάθειας στήριξης μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι λοιπόν σημαντική η ε, διάσκεψη αυτή για την δημοκρατική νομιμότητα. Θα δώσω ιδιαίτερο φως σήμερα σε τρία στοιχεία. Πρώτο, η σημασία του εξαμήνου ως ανταπόκρισή μας στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Δεύτερο, Πώ μπορούμε με τον τρόπο αυτό να προλάβουμε μελλοντικέ κρίσει. Και τρίτο, ορισμένα από τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να μεγιστοποιήσουμε την αξία τη διαδικασία αυτή και σε ό,τι αφορά την τα οικονομικά τη και σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά τη στοιχεία. Πρώτο λοιπόν στοιχείο, ο στόχο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών στα δημοσιονομικά όσο ακόμη προετοιμάζουμε την ανταπόκρισή μας στις διάφορες ελλείψεις ισορροπιών. Τα εξήγησε αυτά ο πρόεδρο Βαν Ρόμποϊ, άρα εγώ μπορώ να προχωρήσω ταχύτερα για να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το εξάμεινο αυτό ήδη από τον Νοέμβριο για να, την έναρξη δηλαδή του 2012 με πέντε προτεραιότητες ενίσχυση της ανάπτυξης αντιμετώπιση της ανεργίας και προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Οι στόχοι αυτοί έχουν ενισχυθεί και από τους ε, αρμόδιους υπουργού στο Συμβούλιο Υπουργών. Την Πέμπτη θα συναντηθούμε εδώ στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί με μένα βέβαια και υπό την Προεδρία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συζητήσουμε τις προκλήσεις αυτές και πώς θα αντιμετωπιστούν. Εκεί θα ανοιχτεί η επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου οι χώρες μέλη θα υποβάλουν τα προγράμματα τους, τα μεταρρυθμιστικά τους δημοσιονομικά προγράμματα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξή. Το εξάμεινο είναι μια διαδικασία αλληλοϋποστήριξης, μάθησης και καθοδήγησης για να εξεύρουμε εφαρμόσιμες στην πράξη λύσεις. Για παράδειγμα, λύσεις όπως η εξής. Για ε, συνεχής καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο, διότι τα προβλήματα είναι κοινά και έχουν κοινέ συνέπειε στο σύνολο δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, διμερείς συναντήσεις με κάθε μια από τις χώρες μέλη που θα ακολουθούνται από στοχευμένε συστάσεις. Επίσης, ομάδε δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, που θα πάνε στις 8 χώρες μέλη που έχουν τα σημαντικότερα προβλήματα ήδη στη διάρκεια του Φεβρουαρίου για να μπορέσουν έτσι να εντοπίσουν του τρόπου με του οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά ταμεία για να προχωρήσει ο κόσμο να βρει δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μονάχα η κλασική μακροοικονομική εποπτεία και ενίσχυση, μπορεί να είναι και ένας πραγματικός διάλογος και μια πραγματική διάδραση για την οικονομική πολιτική και για το πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Εκτός από αυτά, με την διασύνδεση του ε, εξαμήνου και την ένταξή του την ευρύτερη προσπάθεια διακυβέρνηση για την, ε, για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 να παίξουμε ένα ρόλο για να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα. Σταθερότητα που σημαίνει αξιοπιστία. Και δεν θα υπάρξει αξιοπιστία χωρίς ανάπτυξη. Και ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει, δεν, δεν ε, είναι απαραίτητη για να επιληθεί η κρίση. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να μετριάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις πολλών από τις οδυνηρές μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή σε πολλές από τις χώρες μέλη και εκτός από αυτό να επιτευχθεί η κοινωνική αποδοχή αλλά και η πολιτική εφαρμοσιμότητα αυτών των φιλόδοξων προγραμμάτων. Και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι πρέπει να πούμε σαφώς ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη η δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι σημαντικό οι πολίτες της Ευρώπης να αντιληφθούν ποιοι είναι οι στόχοι που επιδιώκουμε με τις μεταρρυθμίσεις αυτές και να κατανοήσουν για ποιο λόγο γίνονται οι θυσίες και ακόμη περισσότερο ότι οι θυσίες αυτές κατανέμονται με δίκαιο τρόπο και δεν επιβαρύνουν μόνο τους ίδιους, τα ίδια μάλλον και πιο τροτά τμήματα της κοινωνίας. Και έρχομαι στο δεύτερο στοιχείο. Πώ μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να αποφευθούν, να προληφθούν κρίσει στο μέλλον. Όλοι αυτοί που αποφασίζουν, οι πολίτε, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι οι οικονομίες μας είναι άρρηκτα συνδεμένες και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκόσμια. Ό,τι συμβαίνει σε μια χώρα μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλες τις άλλες και ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς τι συμβαίνει στην ζώνη ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δείχνει το υψηλό επίπεδο αλληλοδιασύνδεσης της παγκόσμιας οικονομίας. Εμείς φτιάξαμε μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά που είναι από τα σημαντικότερα δυνατά μας σημεία. Και χωρίς αυτήν σίγουρα η κρίση θα είχε πλήξει πολύ βαρύτερα την Ευρώπη. Όμως το σημερινό ανοιχτό οικονομικό μοντέλο, παρόλα του τα πλονεκτήματα απαιτεί και ένα αυξημένο επίπεδο ευθύνης είναι κρίσιμο λοιπόν να βελτιώσουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να αποφευθεί η διασπορά των αρνητικών επιπτώσεων που βλέπουμε στην Ευρώπη από το 2008. Οι δημοσιονομικές αποφάσεις είναι βεβαίως αρμοδιότητα και ευθύνη των εθνικών βουλών και αυτό έτσι θα παραμείνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά βέβαια τι δημοκρατικές διαδικασίες και την διάκριση των εξουσιών. Ο στόχος όμως του εξαμήνου είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου ενδεχόμενες απειλές ή αδυναμίες να μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα με την συλλογή ε, ακριβών πληροφοριών που όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουν να συμβάλλουμε καλύτερα και στην λήψη αποφάσεων και στο εθνικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ισορροπίας καθώς και των επιθύμητων παρενεργειών. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν ανησυχίες και ευαισθησίες όταν, προ... όταν ζητούμε να ανοίξουν τα εθνικά δημοσιονομικά σχέδια στην ευρωπαϊκή εποπτεία. Ωστόσο, αυτοί που κυρίως μας παρακολουθούν είναι εκτός της ενίας αγοράς. Οι παίκτες οι παγκόσμιοι. Λοιπόν, στην ίδια κατεύθυνση κινούμαστε εν τέλει. Το μέλλον μας είναι απόλυτα διασυνδεδεμένο. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σαν εργαλείο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια αύξηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τρίτο, εάν θέλουμε να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Δεν μπορεί να είναι μόνο άνωθεν. Χρειάζεται την στήριξη και την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι επίσης για τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην τελευταία ολομέλεια του Φεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για τη σημαντική, για τη σημαντική σύγκριση των απόψεων των οργάνων μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση σε όλες τις φάσεις του κύκλου. Και αυτό κάναμε προτάσεις τον προηγούμενο Νοέμβριο για να επιτρέψουμε να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια πριν από το Εαρινό Συμβούλιο. Ωστόσο χρειάζονται και διαφορετικά μέτρα επιτόπου για να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Χρειάζονται, γίνονται ήδη σημαντικέ προσπάθειε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικέ μεταρρυθμίσει σε πολλέ χώρε. Ωστόσο, με ανησυχεί η αργή πορεία που σημειώνεται σε, ορισμένες, σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, για τη δημοσιονομική εξυγίανση και πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις ακόμη καθυστερούν Όπω για παράδειγμα στη μεταρρύθμιση των φορολογικών, των συνταξιοδοτικών, τη αγορά εργασία, το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών και τη μεταποίηση. Βέβαια, η εικόνα είναι ανάμεικτη σε όλη την Ευρώπη, όμω αυτή είναι η τομή όπου Κομισιόν και Συμβούλιο ρίχνουν ιδιαίτερο φω στι προτάσει που κάνουν αναχώρα. χώρα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι και δύσκολε και ευαίσθητε. Είναι όμω απόλυτα απαραίτητε για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα. Αναμένω από εσά, την συμβολή σας και τη συνεργασία σας για να γίνει επιτυχία το εξάμεινο. Αναμένω επίσης από εσάς να σφυριλατήσετε τις συνθήκες για να αναπτυχθεί η συζήτηση και η ενημέρωση των πολιτών σας στις χώρες σας. Πιστεύω ότι είναι κρίσιμο για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής, δηλαδή η επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020, η κυριότητα των μεταρρυθμίσεων να παραμείνει στα εθνικά επίπεδα, όχι μόνο στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και στους κοινωνικού εταίρους και στις περιφέρειες. Εδώ χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα, διότι όπως θύμισε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να αποφύγουμε την ιδέα ότι υπάρχει μια αποσύνδεση και καμιά φορά και εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η αποσύνδεση ανάμεσα στα όσα αποφασίζουν εδώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και το τι συμβαίνει μετά στις χώρες μέλη. Καθένα από εμά οφείλει να αναβάλει το ρόλο του για να προωθήσει τη συζήτηση αυτή και να εξηγήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε, να ρίξουμε τα σύνορα και να δείξουμε πώς η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να μας βοηθήσει να φτιάξουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που να στηρίζει την απασχόληση. Και ενώ εδώ κυρίω επενδύσει, θα τα συζητήσουμε και στο στην επόμενη διάσκεψη κορυφή, ιδίω για τα ομόλογα έργων. Θέλουμε να υποβάλουμε προτάσεις και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις επενδύσεις μας, τα διαφθορτικά μας ταμεία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ρίξουμε περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη, ιδίως για παράδειγμα στην υποδομή. Εδώ αλληλοδιασυνδέονται οι μεταφορές, η ενέργεια, τα ε, ψηφιακά. Μιλούμε λοιπόν για μεταρρυθμίσεις, αλλά μιλούμε και για επενδύσεις στο απαραίτητο επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, καθώς και για τρόπους μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων κοινωνικά σε ορισμένων δηλαδή μέτρων που λαμβάνονται. Κυρίε και κύριοι, θα ολοκληρώσω με μια παρατήρηση. Βάζοντας μέσα σε μια διαδικασία όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο συμπεριλαμβάνει και αναπτύσσει το μεγάλο δυναμικό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κλειδί για να ανοίξει το δυναμικό αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία του δυναμικού που έχουμε, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το συνδυασμό του εθνικού επίπεδου, του ευρωπαϊκού επίπεδου, εξασφάλιση της σταθερότητας βραχυπρόθεσμα, αλλά και η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω και μακροπρόθεσμα. Να έρθουν λοιπόν όλα μαζί αυτά τα στοιχεία, η γνώση, τα εργαλεία, θα μας δώσουν τεράστιες δυνατότητες για να προχωρήσουμε σε ανάκαμψη και να αστερώσουμε το μέλλον μας. Αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμός όλων αυτών των εργαλείων και η βέλτιστη δυνατή χρήση τους. Ενίσχυση των συνδέσμων μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών επιπέδων που μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικά ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Έχουμε καθήκον να είμαστε το ίδιο φιλόδοξοι για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας. Η σημερινή συνάντηση μπορεί νομίζω να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την συμμετοχή στη δημοκρατική συζήτηση αλλά και τα απορίσματα των εργασιών σας. Merci Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Και επειδή ο πρόεδρος Βαν θα μας αφήσει σε λίγα λεπτά, θα πρότεινα να ακούσουμε μια πρώτη σειρά τριών ερωτήσεων, στις οποίες θα απαντήσει ο πρόεδρος Βαν και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπους ομιλητές, που είναι αρκετά πολλοί. Ε, και σας ζητώ σε όλους να τηρήσετε πειθαρχία και να μιλήσετε για δύο, maximum τρία λεπτά, για να μπορέσει να γίνει η συζήτηση. Πρώτος έχει ζητήσει το λόγο ο πρόεδρος Μαρίνη, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομίας του Γαλλικής Γερουσίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η συνεδρίαση ίσως να προδιαγράφει την εφαρμογή του άρθρου 13 της μελλοντικής συνθήκης. Θα ήταν δυνατόν να μας πείτε ποια, ποιο όραμα έχετε για αυτές τις περιοδικές συνεδριάσεις. Είναι απλές ενημερωτικές συνεδριάσεις, ε, είναι ένα σώμα καταγραφής γεγονότων, χώρος ε, τεχνικών επαφών, δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας για εμβάθυνση σε διάφορα ζητήματα. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε εν αναμονή τέτοιου είδους διευκρινήσεων. Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για μεθόδους, έννοιες που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, παρατηρούμε όλοι στα εθνικά μας κοινοβούλια ότι αυτές οι ιδέες, αυτές οι έννοιες καθίστανται όλο ένα και πιο περίπλοκες και απαιτούν μακροοικονομική ανάλυση όλο ένα και πιο περίπλοκη και πράγμα το οποίο μας παραπέμπει βέβαια κατανοητό στη δημιουργία ανεξάρτητων δημοσιονομικών επιτροπών στο πλαίσιο των κρατών. Όμως έχω συχνά διερωτηθεί γιατί σε κοινοτικό επίπεδο δεν προβλέπουμε αυτού του είδους την προσέγγιση. Δύο παραδείγματα πριν να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Όσον αφορά το διαρθρωτικό υπόλοιπο που παραπέμπει σε μια αξιολόγηση του, ε, του οικονομικού κύκλου και ε, σημαίνει διορθώσεις. Δεν θα ήμασταν σε καλύτερη θέση και δεν θα δίναμε περισσότερο μια αίσθηση ισότητας αν τα νούμερα δεν θεσπίζονταν μόνο από την ίδια την Επιτροπή, αν υπήρχε μια εξωτερική αντικειμενική γνώμη εμπειρογνωμόνων. Και έπειτα, ακόμα ένα παράδειγμα, η έκθεση της Κομισιόν της 14ης Φεβρουαρίου όσον αφορά το μηχανισμό προειδοποίησης. Όπως και άλλοι παρατήρησα και, και θεωρώ ότι εφόσον πρόκειται για το τρέχον πλεόνασμα, το γεγονός ότι ορίζεται η οροφή στα έξι σημεία του ΑΕΠ, σε έξι ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, αυτό ήταν ε, σκόπιμο, καθώς εξαίρετος εταίρος μας η Γερμανία έχει ακριβώς 5,9 πλεόνασμα σε σχέση με το ΑΕΠ. Είναι κάπως ηρωνική βέβαια η παρατηρήσή μου, αλλά ακριβώς ε, στόχο έχει την αναζήτηση ισότητας και την επιθυμία να έχουμε πιο μακροπρόθεσμα ουδέτερες αναφορές, εμπειρογνωμοσύνες, με τις οποίες να μπορεί κανείς αντικειμενικά να ταυτιστεί και να ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Μαρίνη. Είμαι βέβαιος ότι και οι δύο Πρόεδροι θα θελήσουν να απαντήσουν. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μουριελ Γκέρκενς, που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Βελγικού Κοινοβουλίου. εκφράσω την ε, χαρά μου για την συνεδρίαση αυτή και για την παρουσία του Προέδρου Φανρομποϊ και του Προέδρου Μπαρόζο και ελπίζω πως τα υπορίσματά μας θα αντικατοπριστούν στις επόμενες αποφάσεις. Ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή κυρίως του κυρίου Φαν γιατί πιστεύω πως θα καταλάβει την ερώτησή μου, ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βασίζεται στην οικονομική διακέρνηση, το εξαπλό πακέτο έχει τεθεί σε εφαρμογή και είμαστε υπό διαπραγμάτευση για το, δεύτερο, για το διπλό πακέτο μέτρων. Στην πρόταση κανονισμού που οργανώνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων των δημοσιονομικών, γιατί στα μοσπονδιακά κράτη όπως ε, το Βέλγιο έχουμε προθεσμίες πολύ δύσκολες να τηρήσουμε, διότι πρέπει να ενσωματωθούν στην περίπτωση προσαρμογών που θα χρειαστούν, να γίνουν διαπραγματεύσεις με τις διάφορες ομοσπονδιακές ε, κυβερνήσεις και δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε τέτοιου είδους υποχρέωση. Ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σε αυτό. Και σε σχέση με την προηγούμενη παρέμβαση όσον αφορά την πρώτη έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου για τον μηχανισμό προειδοποίησης που στόχο έχει να εντοπίζει όσο γίνεται πιο γρήγορα τους μακροοικονομικούς κινδύνους στα κράτη-μέλη ε, βρίσκω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αντίθετα με το κανονισμό επί το οποίο βασίζεται αυτή η έκθεση, η Κομισιόν βασίζεται σε μια αντίληψη της ε, σχέσης μεταξύ ανταγωνιστικότητα και κόστο και δεν αναφέρει πότε παράγοντες όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η εξέλιξη του, του ενεργειακού της, της, του ενεργειακού τιμολογίου που είναι πολύ σημαντικό και παίζει τεράστιο ρόλο στα νοικοκυριά. Το ίδιο η απασχόληση και η ανεργία μένουν κατά μέρο. Ενώ το κόστος της ανεργία είναι πολύ υψηλό και γνωρίζουμε ότι η κοινωνική διάσταση μπορεί να είναι πηγή μακροοικονομικής ανισορροπίας. Το ίδιο και για τα ποσοστά φτώχειας. Και έπειτα, ως, βουλευτές, ως βουλευτής λυπούμε που αν και βρίσκεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να εξετάσει τα σημαντικά πλεονάσματα όσον αφορά τις χώρες μάλλον που έχουν σημαντικά πλεονάσματα στο εμπορικό τους ισοζύγιο και ασχολείται μόνο με συγκεκριμένες χώρες και χώρες που θεωρούνται υπεύθυνε για την κρίση λόγω της ε, μισθολογικής μετριοπάθειας που, τηρεί, που τηρούν. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για την ε, έννοια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία έχει όμως ε, μετατραπεί. Αρχικά επρόκειτο για μια ετήσια εξέταση για την ανάπτυξη που βασιζόταν στη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αυτή η στρατηγική έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορες πρωτοβουλίες ε, πολύ σημαντικές και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν υπάρχουν πια αυτέ οι πρωτοβουλίε. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι κατευθυντήρες γραμμέ οι δείκτες, για τι βιομηχανικέ, πολιτικέ, σε εθνικό επίπεδο και εδώ δεν γίνεται καν λόγο για αυτά, ούτε στο ενετήσια εξέταση για την ανάπτυξη. Το ίδιο και στο φύλλο πορεία για μια αποτελεσματική Ευρώπη στη χρήση των πόρων. Εντάχθηκε αυτό στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από φέτο και στο εξή και εδώ και πάλι δεν βλέπουμε να γίνεται μια υλοποίηση. Το ίδιο και για άλλες πρωτοβουλίες όπως η καταπολέμηση της ένδυα, η πρόσβαση στην παιδεία και ούτω καθεξής. Αυτή η εξέλιξη νομίζω πως είναι ανησυχητική εάν θέλουμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση που θα επιτρέπει να λαμβάνονται μέτρα ανάπτυξης χωρίς να πέσουμε σε μια λιτότητα η οποία τελικά θα είναι στήρα όσον αφορά την ε, εξέλιξη μια εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή πολιτική. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τελευταίο ο μιλητής είναι ο Σαλβατόρ Γκαρίγκα από την Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια διαφορετική διάσταση γιατί άλλωστε είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ιδέα του εξαμήνου αυτού ως προς την ε, υποβολή των εθνικών προϋπολογισμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την ε, δική μας Επιτροπή. Ωστόσο, ελάχιστη είναι η σχέση μεταξύ εθνικών προϋπολογισμών και κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αυτό ο συντονισμός. Το 80% ε, δαπανάται και τροφοδοτούμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό με εθνικές συνεισφορές που πρέπει να εγκρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ο προϋπολογιστικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και ολοκληρώνεται το Νοέμβριο με τη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Είναι δύσκολο να βρεθεί ένα καλύτερο όχημα συντονισμού μεταξύ 27 εθνικών προϋπολογισμών και τον 28ο προϋπολογισμό που είναι ο κοινοτικό προϋπολογισμός. Είναι πιο δύσκολο λοιπόν να βρεθεί όχημα, όχημα καλύτερο από το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εξού λοιπόν και έχουμε ε, καθορίσει όλα αυτά τα κριτήρια και το βασικό κριτήριο είναι να έχει κάτι ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ως εκ τούτου, αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στον Πρόεδρο Φαν Ρομπό και στον Πρόεδρο Μπαρόζο είναι το εξή. Να χρησιμεύσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ούτως ώστε να αντικατοπτριστούν στον κοινοτικό προπολογισμό οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των Εθνικών κοινοτικών προπολογισμών και αντιστρόφως. Εμείς δηλαδή στον δικό μα κοινοτικό προπολογισμό, να είμαστε σε θέση να αντικατοπτρίσουμε τι ευαισθησίε που θα εγκρίνουν ή που έχουν εγκρίνει τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φαν Ρομπόη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τις ε, ερωτήσεις που μου τέθηκαν, ωστόσο είναι αρκετά εύκολο το εγχείρημά μου διότι ή θα πρέπει να αναφερθώ στο διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ε, θα αφήσω το λόγο να το πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν έχω, ξέρετε, πάντοτε εύκολα εγχειρήματα να φέρω σε, πέρος, σε πέρας. Όμως ε, με αυτές τις τρεις πρώτες ερωτήσεις νομίζω ότι είναι εύκολο το καθήκον μου να κάνω κάποια προκαταρκτικά σχόλια. Το άρθρο 13 της νέας συνθήκης, στο οποίο αναφερθήκατε ε, και το οποίο ε, ε, πρέπει να κυρωθεί, αφήνει απολύτως ανοιχτό τον τρόπο με τον οποίο θα διοργανώσουν τις διαβουλεύσεις τους τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό έχει γίνει εσκεμένα ή θελημένα. Δεν θέλαμε εμείς ως ε, όλοι όσοι διατύπωσαν το κείμενο της συνθήκης να ε, προσδιορίσουμε επακριβώς τις ε, εφαρμοστικές λεπτομέρειες με τις οποίες θα λάβει η χώρα αυτή η διαβούλευση και αυτή η συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές όμως ότι αναφερόμαστε σε αυτή τη συνεργασία ε, και σε αυτή την αλληλεξάρτηση και αυτό είναι ένα πολιτικό γεγονός καθεαυτό. αυτό. Εσείς πλέον μετά ε, πρέπει να αναλάβετε την, αυθή, την ευθύνη να οργανώσετε τις εργασίες σας με τον, ε, όσον τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ούτως ώστε να συμβάλλουν όλοι ε, όσο περισσότερο μπορούν. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Μία δεύτερη παρατήρηση ως προς τις ανεξάρτητες φωνές, τους αυτόνομους, τους ανεξάρτητους και τη συμβολή τους στην υλοποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων. Βεβαίω θα πάρει το λόγο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εργάζεται εν κενό. Όταν για παράδειγμα προσπαθεί να δώσει τον ορισμό ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, ε, αυτόν τον ορισμό τον δίνει έχοντας ακούσει, έχοντας διαβάσει, έχοντας μελετήσει όλα ε, τα πορίσματα και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα ως προς αυτή την τόσο περίπλοκη έννοια. Επομένως κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει σε μια συγκεκριμένη πρόταση είναι πάντοτε τεκμηριωμένη η πρότασή της και στηρίζεται στην διαφάνεια, στις αρχές της διαφάνειας, της διαφάνειας και ε, στην επιθυμία να ε, καταστήσει τα πάντα πιο προσβάσιμα σε όλους και γι' αυτό πάντοτε δίνει τους σωστούς ορισμούς ε, στις μεθόδους και στα νοήματα τα οποία προβάλλει. Εάν δεν ανατεθεί αυτό το καθήκον σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι το μόνο που θα κάνουμε είναι να χρονοτριβούμε ε, με άσκοπες συζητήσεις. Για εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, το οποίο βεβαίως συνεργάζεται στενά με πάρα πολλά ερευνητικά ιδρύματα, ε, καταλήγει σε έναν ορισμό και εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον ορισμό. Ως προς την χρονική συγκυρία, να πω στην Βελγίδα συνάδελφο ότι βεβαίως το Βέλγιο είναι μια πολύ περίπλοκη χώρα, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν είναι μόνη. Δεν είναι και η μόνη. Υπάρχουν πολλά ομοσπονδιακά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ισπανία ενδεχομένω και σε μικρότερο βαθμό και άλλες χώρες θα έλεγα. Επομένως η χρονική συγκυρία είναι μια συνολική συγκυρία αυτό το οποίο αποκαλούμε timing δηλαδή. Ωστόσο, ε, φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εξαιρετικά νωρίς με την ετήσια μελέτη ε, για θέματα ανάπτυξης. Το Annual Growth Survey το ξεκίνησε και το παρουσίασε τον Νοέμβριο από την προηγούμενη χρονιά. Γνωρίζω ότι σε ορισμένες χώρες προέκυψε κυβέρνηση εξαιρετικά αργά Άλλο θέμα αυτό βέβαια. Αλλά σε ένα φυσιολογικό κύκλο ε, εξελίξεων νομίζω ότι μπορεί να οργανωθεί κανείς ούτως ώστε να υπάρχουν από τον Απρίλιο ε, τα σχέδια μεταρρύθμισης και τα σχέδια σταθερότητας. Ακόμα και σε χώρες που έχουν μια διοικητική διάρθρωση αρκετά περίπλοκη και αρκετά ομοσπονδιακή. Τρίτη παρατήρηση ε, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα. Είναι βεβαίως πάντοτε πολύ λεπτή αυτή η επιλογή ποιος είναι ο σωστός δείκτης. Μια χώρα την οποία γνωρίζετε και την οποία εγώ γνωρίζω καλύτερα από άλλους, έχει ένα δίκτυο ανταγωνιστικότητας και η παράμετρος αυτή είναι η παράμετρος την οποία ε, θέσαμε ενώπαιόν σας και η παράμετρος ε, την οποία ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι βέβαια η μόνη παράμετρος αυτή. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου γίνεται λόγος για προβλήματα ανταγωνιστικότητας, τα οποία όμως ε, δεν εστιάζονται αποκλειστικά και μόνο στους μισθούς. Ε, θα... Δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένη χώρα, αναφέρω όμως μια χώρα η οποία δεν είναι και η χειρότερη άλλωστε, ε, στην οποία αναφέρεται έλλειμμα και μείωση ανταγωνιστικότητας λόγω μείωσης και ελλείμματος καινοτομία. Δηλαδή η έννοια της ανταγωνιστικότητας βεβαίως περιλαμβάνεται στους δείκτες ε, και έχουμε τον πολύ γνωστό ε, δείκτη ε, που έχει συμπεριληφθεί και στη βελγική νομοθεσία. Συνολικά όμως, όταν αξιολαγούνται οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, η παροχή των υπηρεσιών και του καθεξής, λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία πολύ πιο ποιοτικά ε, και δεν λαμβάνεται μόνο υπόψη η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο κόστους, αλλά και η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο ε, προϊόντων. Αυτές είναι κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις ως προς τις ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ως προς το τελευταίο ερώτημα, παρόλο που και αυτό ε, εντάσσεται περισσότερο στο ε, πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι προϋπολογισμοί των ΜΕΝ και των ΔΕ είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να σας το εξηγήσει καλύτερα πολύ καλύτερα από ότι εγώ. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας προϋπολογισμός επενδύσεων σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίω, στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων είναι πολύ μεγάλη η συνεισφορά των κρατών μελών. Και άλλωστε κάποια κράτη-μέλη παραπονιούνται γιατί θεωρούν ότι εισφέρουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν όλα αυτά έχοντα δική μα φορολόγηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι προπολογισμό δαπανών, είναι προπολογισμό επένδυση κατά κύριο λόγο. Ενώ οι εθνικοί προπολογισμοί έχουν μια τελείω διαφορετική φύση. Το 40 ή το 50% του προϋπολογισμού σε ορισμένες χώρες αφορά δαπάνες ε, κατανάλωσης ή ε, μεταφορών, ε, μετακύλησης. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά τα δύο εγχειρήματα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Και μάλιστα διαφέρονται και ως προς τον όγκο τους. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει να κάνει με το 1% του, του ευρωπαϊκού προϊόντος, του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αν θέλετε, ενώ ο προϋπολογισμός μιας χώρας μπορεί να φτάσει στο 50% του εγχώριου του ΑΕΠ της χώρας αυτής. Βλέπετε πόσο ε, μεγάλη είναι η διαφορά ως προς το ποσοτικό βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εθνικών ε, προϋπολογισμών. Ωστόσο και σε ποιοτικό επίπεδο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι τελείως διαφορετικής φύσης αν θέλετε. Επομένως είναι λιγότερο σημαντικό να προσαρμοστούν τα χρονοδιαγράμματα από τη στιγμή που το εχείρημα αυτό διαφέρει ε, ιδιαιτέρως ε, Ω προ του εθνικού προϋπολογισμούς από τη μία και τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό από την άλλη. Αυτές είναι κάποιε προκαταρκτικές παρατηρήσεις που θα μπορούσα να κάνω. Να επαναλάβω όμως ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περισσότερο αρμόδιος για να απαντήσει ε, συγκεκριμένα σε αυτές τις τρει ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και για τις απαντήσεις σας. Σας προτείνω να συνεχίσουμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις και ο πρόεδρος Μπαρόζο θα απαντήσει μαδικά στο τέλος σε όλους. Μπορείτε να συνεχίσετε λοιπόν, να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας, έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι να πάρουν το λόγο. Δίνω το λόγο στο πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών του Λέντους Κούντακτ της Φιλανδίας, το Κίμους Χασί. Συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν θεσπίστηκε το ευρώ και υπογράφηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όλοι γνώριζαν ότι ήταν πολύ σημαντικό η συμφωνία αυτή να τηρηθεί. Ξέραμε όλοι ότι αν δεν το θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Δεν τηρήθηκε ωστόσο και γι' αυτό ξέσπασε η κρίση χρέους, γι' αυτό το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το να μην τηρηθεί αυτό το σύμφωνο σημαίνει ότι δεν τηρούμε απόλυτα το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Κομισιόν έρχεται με το εξαπλό πακέτο, το διπλό πακέτο, το δημοσιονομικό πλαίσιο, την πειθαρχία κτλ. Είναι καλές οι προτάσεις αυτές καθ' αυτές, ωστόσο είναι πολύ περίπλοκες και μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα για ένα-δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα όταν οι αγορές λαμβάνουν αποφάσεις σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλοί και αποτελεσματικοί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα ήταν δυνατόν, γιατί πολλές χώρες θέλουν να μπουν στο ευρώ. Αν όμως επί τρία χρόνια ε, παραβιάζεται το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη ότι θα βγαίνει κανεί από το ευρώ και έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα σύγκρουση. Αν μια χώρα μέσα σε τρία χρόνια δεν μπορεί να τηρήσει το σύμφωνο σταθερότητα και ε, ανάπτυξης ε, να βγαίνει από το ευρώ. Πολλέ χώρε θέλουν να μπουν στο ευρώ, αλλά πολύ λίγε θέλουν να βγουν από το ευρώ. Είναι καλή αυτή η πρόταση, θα τη στηρίζατε εσεί. Σα ευχαριστώ για αυτέ τι ε, προκλητικέ ιδέε, αλλά οφείλουμε, οφείλουμε να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος, από όλες τις χώρες μέλη του ευρώ, η Φιλανδία είναι η μόνη που έχει τηρήσει όλα τα κριτήρια σωστής, ορθής διαχείρισης εξ αρχής. Ο πρόεδρος Μπαρόζο λέει ότι ακόμα και η Φιλανδία παραβίασε για κάποιο μικρό διάστημα το σύμφωνο αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Παίρνουμε στη Σκανδιναβία με τους καλούς μαθητές, αλλά αφήνουμε την Ευρωζώνη για την ώρα και δίνουμε το λόγο σε έναν εκπρόσωπο του Ρικ Στάγγεν της Σουηδίας, την κυρία Ελίζαμπετ Σβάνσον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσε τις σημαντικές αυτές συζητήσεις. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη γνώμη σας σχετικά με την κρίση εμπιστοσύνης σε από πολλές πτυχές οφείλεται βέβαια στην κρίση χρέους, αλλά είναι και κρίση αξιοπιστίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μας και πάνω της, της, αξιοπιστίας μας μάλλον και της εμπιστοσύνης των αγορών την εμπιστοσύνη αυτή θα την επιτύχουμε μονάχα εάν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα όσα έχουμε αποφασίσει. Για παράδειγμα, τα μέτρα της ε, δέσμης των έξι οδηγιών ή των δύο οδηγιών. Α, πρέπει να αποκαταστήσουμε υγιή δημοσιονομικά σε όλες τις χώρες μας. Και αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει με ταυτόχρονο σεβασμό της κυριαρχίας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όλοι επιθυμούμε μεγαλύτερη και περισσότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Βεβαίω και πρέπει να έχουμε στραμμένα τα βλέμματα στο μέλλον, αλλά μας ανησυχεί όταν ακούμε εδώ διαρκώς για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που υποτίθεται ότι θα προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει μονάχα όταν βασίζεται σε μια η υγιή οικονομία. Όταν υπάρχουν πληγές που ματώνουν, πρέπει πρώτα αυτές να επουλωθούν. Αυτό ισχύει και για τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις είναι σκληρές, πονούν, αλλά αυτές είναι που πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν και μετά μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη πρέπει πρωτίστως να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Εκεί υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν άλλου είδου επεκτατικά μέτρα. Αυτό που χρειάζεται είναι να λειτουργήσει η ενιαία αγορά. Χρειάζεται να φροντίσουμε ώστε να εξηγιανθούν τα δημοσιονομικά και μετά θα πετύχουμε και την ανάπτυξη. Αυτό θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Κυρία μου, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αλεχάντρο Σέρκας, μέλος της Επιτροπής Απασχολήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος ε, της ομάδας των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την απασχόληση και τα εργασιακά θέματα σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και πώς θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε μια μεσομακροπρόθεσμη ε, οπτική γωνία σε ένα εγχείρημα το οποίο αν δεν την αποκτήσει αυτή τη διάσταση θα απέχει πόρο από τις ε, ε, προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, κύριε Φαν Ρομποέ, ως Ευρωπαίος πολίτης, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι οι σχηματισμοί του Συμβουλίου ε, δίνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος στις οικονομικές διαστάσεις παρά στις ανθρώπινες ή εργασιακές. Ελπίζουμε ε, στη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Άνοιξης να διαβάσετε ε, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πυλώνων. Άλλωστε η οικονομία ή θα εξυπηρετήσει, θα στηρίξει και θα βοηθήσει ούτως ώστε ο ανθρώπινος παράγοντα να προορέσει να ευημερήσει και κυρίως η νέα γενιά ή αλλιώς δεν έχει και μεγάλη χρησιμότητα αν θέλετε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία θέλει να ακουστεί η φωνή του στην νεαρινή σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ούτω ώστε να εξεταστεί το δράμα που βιώνει η νέα γενιά στην Ευρώπη, το ε, δράμα της ανεργίας γενικότερα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξει το, η Σύνοδος τόσο πολύ όσο προσέχει ε, και το θέμα των, ε, του εθνικού χρέους ή όλης της οικονομικής κρίσης. Έχουμε εκατομμύρια νέους που αναζητούν δουλειά και αναζητούν αν θέλετε και μια ακτίνα ελπίδας και εκατομμύρια ανθρώπους που ε, βρίσκονται στο χείλο της φτώχειας ή έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας. Ζητούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να μην παραγνωρίσει ε, τη βασική στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Να μην λειτουργήσουμε μόνο βραχυπρόθεσμα. Εάν η Ευρώπη δεν έχει τη φιλοδοξία να κερδίσει το παιχνίδι σε βάθος χρόνου, να δημιουργήσει πραγματικά ουσιαστική απασχόληση, όχι οποιαδήποτε απασχόληση, αλλά απασχόληση που θα επιτρέψει την επίτευξη της υπεροχής. Μόνο έτσι ε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο William Cash της ε, ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Βουλής των Κοινοτήτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εκφραστώ ελεύθερα και να εκφράσω την άποψή μου σε αυτή την συνάντηση σήμερα και θα το πράξω και μάλιστα με πολύ μεγάλη ε, συντομία. Ε, άκουσα τον κύριο Φαν και τον κύριο Παρόσο να μιλούν για τη δημοκρατία. Τους άκουσα να μιλούν για τη δημοκρατική νομιμότητα. Οφείλω να πω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία εμείς στο Κοινοβούλιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Η συνθήκη των 25 Από τα στοιχεία που έχω λάβει από την έρευνα που διεξάγουμε στη Βουλή των Κοινοτήτων για αυτό το θέμα, ε, τελεί ε, ε, επιπαραβάση όσον αφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Και όταν ακούω ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σύμφωνα με τον κύριο Φαν Ρομπάι, αυτό δεν ισχύει θέματα που έχουν να κάνουν με φορολόγηση και δαπάνες ε, είναι θέματα εθνικών κοινοβουλίων που αποφασίζονται ε, από εκλεγμένους, από τον λαό. Δεν μπορείτε συνεχώς να λέτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και περισσότερη Ευρώπη, ως να είναι αυτό ε, ένα οσανάτο που θα πρέπει να αναφωνήσουμε όλοι από κοινού. Τα αληθινά προβλήματα έγκυται στην έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας, στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας και στο έλλειμμα σεβασμού των αποφάσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και θέλω μάλιστα ε, να καταλήξω κάπου εδώ λέγοντας ότι το θέμα εθνικής ταυτότητας και εθνικής λήψης αποφάσεων ε, δεν είναι ένα θέμα αφηρημένης, ε, αν θέλετε, ιδεολογίας. Είναι θέμα καθημερινής ελευθερίας, πολύ συγκεκριμένη. Ελευθερίας ψηφοφόρων να αποφασίζουν οι ίδιοι τι είδους κυβέρνηση και ποια είδους κυβέρνηση θέλουν. Όταν μιλούμε για όλο και περισσότερο η Ευρώπη, αυτό ενδεχομένως αυτό είναι η αιτία του προβλήματος και το λέω ως κάποιος του οποίου ο πατέρας πέθανε στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο πολεμώντας για την ελευθερία. Εμείς πιστεύουμε στην ελευθερία που εκπορεύεται από τον ατομικό ψηφοφόρο ο οποίος εκφράζει την άποψή του στις γενικές εκλογές. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Και η αιτία του προβλήματος, την οποία δεν αναγνωρίζει και κανείς, είναι ότι αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, ούτως ώστε να, να κατοχυρωθεί αυτή η αρχική αξία της ελευθερίας, ούτως ώστε να ξαναποκτήσουμε τη, τη δημοκρατία την οποία ε, πήραν από τα χέρια μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας απαντήσει επί της ουσίας ο πρόεδρος Μπαρόσο. Νομίζω όμως ότι χαίρεστε, είστε ικανοποιημένος, διότι συμμετέχετε σε μια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν μόνο αιρετοί δημοκρατικώς εκλεγμένοι ε, ηθήνοντες. Και δυστυχώς η η προσωπική σας τραγωδία σχετικά με το θάνατο του πατέρα σας είναι ε, μια τραγωδία η οποία αγγίζει όλους εμάς. Ο καθένας από εμά έχει γονείς που έχουν χάσει τη ζωή τους στον τελευταίο ε, πόλεμο. Εξού και βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αλευρά. Thank you, ε, I would like to, some remarks. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Δεν έχω αντίρρηση. Καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίρρηση κατά των κυρίων στόχων του νέου συμφώνου. Καταλαβαίνω πως είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις Ευρω... χώρες του Ευρωζώνη να καταπολεμήσουν το έλλειμμα και το χρέος. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχουμε ενώπιον μας ένα νέο σχέδιο που δεν είναι πολύ δημοφιλές και δεν θα μπορούσε να είναι πολύ δημοφιλές. Διότι σε αυτή την περίοδο πρέπει να καταπολεμήσουμε το χρέος, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την ύφωση. Στι πολλέ νότιε χώρε αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρή ύφεση που καταστρέφει τη ζωή των ανθρώπων και δεν έχουμε βρει λύσει. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα, το κύριο θέμα σε σχέση με αυτή την στρατηγική Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ώστε αυτό το σχέδιο τελικά δεν είναι πολύ ε, δημοφιλέ. Είναι καλό τεχνικό σχέδιο, αλλά δεν έχει πολιτική υφή. Και δεν θα μπορούσε να είναι πολιτικό σχέδιο αν οι Γερμανοί είναι πάντοτε υπό την πίεση να πληρώνουν περισσότερα και οι Έλληνε είναι πάντοτε ανήσυχοι για να κάνουν περισσότερα, για να δεχτούν κάποια, να μπορέσουν να έχουν κάποια οικονομική βοήθεια. Καταλαβαίνω πως ε, χρειαζόμαστε αυτού του είδους ε, την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά δεν δίνεται καμία απάντηση στο πώς θα συντηρήσουμε το κοινωνικό κράτο, την κοινωνική προστασία, την κοινωνική πρόνοια. Δεν έχουμε κοινέ προδιαγραφέ για την κοινωνική πρόνοια στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πρόβλημα. Ε, νομίζω πω χρειαζόμαστε κάποιε κοινέ αρχέ, κάποιε κοινέ προδιαγραφέ για την κοινωνική πρόνοια στην Ευρωζώνη. Γιατί χωρί κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε βιώσιμε λύσει στου λαού μα, Ευχαριστώ. Ε, je donne la parole à M. Kleina, représentant le Sénat de Pologne κ. Κλεινά της Πολωνικής Γερουσίας. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριε και κύριοι, η Πολωνία έκλεισε τον περσινό χρόνο με πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα. Με 4% οικονομική ανάπτυξη. Φέτος αναμένουμε πάλι θετικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και μεταρρυθμίσεις για δημοσιονομικά και για το συνταξιδοτικό μας, διότι θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να γίνουν, διότι έχουμε καλή οικονομική ανάπτυξη και διότι στη βάση αυτή θέλουμε να προλάβουμε μελλοντικές κρίσεις. Υποστηρίζουμε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα βελτιώσει την οικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό στα δημοσιονομικά. Γνωρίζουμε ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη. Με συναντήσεις όπως η σημερινή θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωρών μας. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο καθιστά ευχερέστερο για τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή συζήτηση. Ήδη σε πρώιμη φάση των εργασιών. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι θετικό, διότι οι εθνικές βουλές είναι αυτές βέβαια που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Πρέπει να εξεύρουμε μια ισορροπία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα είπαν αυτά και άλλοι συναδελφοί μου πριν, και ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός πρέπει να μπορέσει να εξηγιανθεί. Έσοδα και δαπάνες πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Υπάρχει μια φυσική τάση να δαπανούμε και όλο και περισσότερο, αλλά αυτή πρέπει να την ελέγξουμε. Οι συστάσεις προς τις χώρες μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα δύο αυτά στοιχεία και όπως είπα να εξεύρουν μια θέση ισορροπίας ανάμεσά τους. Όπως είπα η χώρα μου, η Πολωνία, επιβάλλει τώρα, αποφασίζει, εγκρίνει και επιβάλλει δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και η ταχύτητα της δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι πολύ σημαντική. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να έχουμε μειωμένα φορολογικά έσοδα. Γι' αυτό τα μέτρα μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στοχευμένα και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας μέλους. Εν αυτών των γεγονότων, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε βέβαια ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση για όλες τις χώρες, κοινή δηλαδή για όλες τις χώρες. Το κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας μέλους. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή δημοσιονομικών βασικών αρχών που θα διασφαλίζουν ότι κάθε χώρα μέλος έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους μηχανισμούς για να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Χρειάζεται διακυβέρνηση και εποπτεία. Χρειάζεται πρόληψη. Η Πολωνία πιστεύει ότι με τα μέτρα αυτά έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε μελλοντικέ κρίσεις καθώς επίσης και περισσότερες δυνατότητες να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Η Πολωνία βρίσκεται εκτός της ζώνης ευρώ. Ωστόσο, οι επιπτώσεις από τις διαταραχές που σημειώνονται μέσα στην Ευρωζώνη φτάνουν μέχρι σε εμά. Γι' αυτό και χρειάζονται μέτρα για τα δημοσιονομικά, τα οποία θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον και το δικό μας. Ο κ. Οκνοκ μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις χώρες όπου τα πειράματα δημοσιονομικής εξυγένσης επέτυχαν, αυτές οι χώρες δεν μπορούν να προσαρμόσουν τις ισοτιμίες τους. Ξέρουμε ότι στις χώρες τη Ευρωζώνης αυτή η προσαρμογή είναι αδύνατη διότι έχουμε το κοινό ενιαίο νόμισμα και υπό αυτές τις συνθήκες οι πολιτικές διαρθρωτικής προσαρμογής κινδυνεύουν να καταλήξουν σε ένα παιχνίδι αρνητικό ή μηδενικό. Γιατί αν όλες οι χώρες μειώσουν τους μισθούς τους ταυτόχρονα, η εσωτερική ζήτηση στην Ευρώπη θα πληγεί και χωρίς ζήτηση οι ίδιες οι επενδύσεις μέσω μιας αντίθετης επιτάχυνσης ε, θα ε, ζημιωθούν. Ξέρουμε όμως ότι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας κυρίως παίζεται στο πεδίο των επενδύσεων και υπ' αυτές τι συνθήκε οι δημοσιονομικές πολιτικές μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο αν δεν γίνεται αν αποτύχει η προσαρμογή των ισοτιμιών ή του ε, κόστους ε, του μισθολογικού. Όμως σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι όπως ε, με αυτά που προτείνει μπορεί να πιέσει πολύ τις νομισματικές πολιτικές. Ο κύριος Βανερομπόη μας θύμισε πριν από λίγο πως έχουμε ένα πραγματικό επενδυτικό προϋπολογισμό μάλλον επενδύσεων που περιορίζεται σε λιγότερο από το 21% του κοινοτικού ΑΕΠ αν ο προϋπολογισμός επενδύσεων των βασικών χωρών της Ευρωζώνης ανέρχεται ανάλογα με την χρονιά ε, στο 3 με 4% ε, του ΑΕΠ των χωρών αυτών. Μιλώ για τον προπολογισμό επενδύσεων. Και ειδού η ερώτησή μου. Σας ε, ζητώ να το σκεφτείτε σε κάποιο καιρό όταν η Ευρώπη θα είναι σε ύφεση, γιατί προβλέπετε ότι το επόμενο χρόνο ο επόμενος χρόνος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος από συγκυριακή άποψη για την Ευρωζώνη. Υπ' αυτέ τις συνθήκες λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε αυτή την πρόταση που έχουμε κάνει κάποιοι από εμά, να αποκλείσουμε από τον υπολογισμό των εθνικών ελλημάτων αυτές τις δαπάνες επενδύσεων για να μπορέσουμε να φτάσουμε από κοινού το στόχο της ε, διαχείρισης των δαπανών και την ανάκαμψη και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, έχετε πολλά να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Θα βλέπω πως όχι μόνο έχω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντί μου, αλλά και το προνόμιο να έχω και τα εθνικά κοινοβούλια απέναντί μου. Και αυτό είναι με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί εγώ εξελέγην ε, σε ηλικία 29 ετών στο Εθνικό Κοινοβούλιο και έκτοτε εκλέγομαι σε όλες τις ε, εθνικές εκλογές και γι' αυτό και μου αρέσει πολύ ο πολιτικός λόγος και η πολιτική συζήτηση. Ο πρόεδρος Φανροπόη νομίζω ήδη απάντησε, αλλά ήθελα και εγώ να κάνω το σχόλιο μου στην κυρία Κέρκενς ε, που αναφέρθηκε σε ορισμένες πτυχές πολύ σημαντικές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα περιλαμβάνονται στις συστάσεις μας αναχώρα Κάθε φορά που κάνουμε μια ανάλυση για την ανάπτυξη, την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη, δεν επαναλαμβάνουμε όλο τον κατάλογο των μέτρων για τη στρατηγική 2020. Ο κ. Σέρκα είπε και σωστά πω υπάρχει μια στρατηγική για την ανάπτυξη. Είναι στρατηγική 2020. Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά που εκδίδουμε ένα νέο έγγραφο τη Επιτροπή να επαναλαμβάνουμε ολόκληρο τον κατάλογο. Και τα όσα είπατε για τη σημασία τη έρευνα και τη ανάπτυξη, για τη βιομηχανία, για την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, των πόρων, το θέμα της καταπολέμησης της ένδυας. Ακριβώς αυτά έχουμε εντάξει στη στρατηγική 2020 και μάλιστα με πολύ μεγάλη δυσκολία σε ορισμένες περιπτώσεις, ε, γιατί εφόσον βρισκόμαστε σε πολιτική συζήτηση θα το πω, πολλές κυβερνήσεις έλεγαν ποτέ δεν πρόκειται να δεχτούμε να μπουν τέτοιου είδους στόχοι όπως η καταπολέμηση της ένδυας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι λόγω της αρχής της επικουρικότητας δεν έχει καμιά δουλειά η Ευρώπη να ανακατεύεται στην καταπολέμηση της στόχης. Αυτό είναι πολιτικές ε, εθνικές. Εγώ χρειάστηκε να αγωνιστώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να πετύχω τη συνένεση στο τέλος, ότι ανάμεσα δηλαδή στους στόχους της στρατηγικής 2020 να είναι και αυτός ο στόχος της καταπολέμησης ένδυα, πέρα από την έρευνα και την ανάπτυξη και τους υπόλοιπου στόχου. Αυτά τα λέω για να σας δείξω σαφώς ότι η στρατηγική 2020 με τις ναυαρχίδες της, όλα αυτά τα προγράμματα που δεν επαναλαμβάνουμε τακτικά, είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Τώρα, στην ετήσια έκθεση ανάπτυξης, είναι αλήθεια, εστιάσαμε την προσοχή σε ορισμένες πτυχές. Όμως τώρα είμαστε μέσα στη διαδικασία διαλόγου με τα κρατημέλη και στη συνέχεια θα διατυπώσουμε τις συστάσεις μας σε εθνικό επίπεδο. Και είμαι βέβαιος πως αυτές οι ανησυχίες που εκφράσατε θα καλυφθούν σχεδόν όλες. Και μάλιστα το σημαντικό ζήτημα της βιομηχανία λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και μάλιστα όταν μιλάμε για το κόστος παραγωγής, όταν μιλάμε για το ποσοστό κάθε κράτους μέλους στις εξαγωγές της Ένωσης και επίσης για το πώς ε, προχωρά η πίστοση για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά όλα συμπεριλαμβάνονται στο θέμα της αντιμετώπισης ε, του κράχ των πιστώσεων, ε, της πίστοσης. Ε, τώρα, για τον κύριο Μαρίνη, μίλησε για σημαντικά θέματα. Το έχουμε συζητήσει επί μακρόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με τα κράτη της ζώνης ε, του ευρώ. Σε ποιον αναθέσουμε αυτό το καθήκον, το αναλυτικό, το υποπτικό, και αυτό της εφαρμογής και το συμπέρασμα που νομίζω είναι δίκαιο είναι να το, να το αναθέσουν στην Κομισιόν γιατί εξορισμού είναι αναξάρτητοι από τα κράτη-μέλη. Εάν τώρα κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα να δημιουργούμε ένα νέο θεσμικό όργανο, ένα άλλο θεσμό, Ορισμένοι θα πούνε και δικαίω που το σύστημά μας είναι ήδη περίπλοκο, θα, θα έχουμε ένα σύστημα τελείως ε, δυσανάγνωστο στο τέλος. Η Κομισιόν λοιπόν είναι το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που έχει αυτό το έργο με βάση τη συνθήκη. Αυτό που ζητώ λοιπόν είναι από όλου του εθνικού βουλευτέ είναι να τηρήσουν τα θεσμικά όργανα που τα κράτη-μέλη ασκώντα τι εξουσίε του, έχουν καθορίσει τα ίδια ω θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιουργήθηκε από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το που είναι άμεσα εκλεγμένο και με πλήρη δημοκρατική νομιμότητα και θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε λίγο. Γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τράπεζα που είναι ανεξάρτητη. Γι' αυτό Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επίσης ανεξάρτητο όργανο. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι, και σίγουρα δεν μιλώ για σας, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω πως ορισμένοι δεν θέλουν αυτά τα ανεξάρτητα όργανα και θέλουν να δημιουργήσουν άλλα θεσμικά όργανα παράλληλα που τι θα κάνουν, θα θα θέσουν σε, θα, θα δημιουργήσουν ανομία όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και θα δημιουργήσουν ακόμη πιο περίπλοκο χαρακτήρα. Δουλέψουμε λοιπόν με τα θεσμικά όργανα που υπάρχουν με σεβασμό στα εθνικά ε, θεσμικά όργανα που έχουν δημοκρατική νομιμότητα αλλά και με τα ευρωπαϊκά όργανα που έχουν δημιουργηθεί όλα μέσω συνθήκων με ομόφωνες αποφάσεις και εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τις αρχές της αντιπροσωπευτικής ε, δημοκρατίας. Τώρα, να τα πω τώρα στα αγγλικά. Ο φίλος μας από την Φιλανδία έκανε μια πολύ προκλητική ερώτηση, όπως είπε και ο φίλος μου Λαμασούρ, μετά από τρία χρόνια έξω από το ευρώ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω πως ε, αυτό είναι η σημερινή συζήτηση. Τώρα μόλις τα κράτη-μέλη, όπως ξέρετε, ενέκριναν δεν, ήταν καν, ε, δεν μπόρεσαν να το εγκρίνουν τα 27 κράτη-μέλη, αλλά ενέκριναν ε, το fiscal compact που είναι μια συνθήκη με σαφείς κανόνες για την Ευρωζώνη. Και όχι μόνο για τα 17 μέλη του Ευρωζώνης, αλλά σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από ένα-δυο, αποφάσισαν να υπογράψουν αυτούς τους κανόνες. Και Η, σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες, τις ισχύουσες συνθήκες δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Είμαστε βέβαια σε μια ομάδα προβληματισμού, το, κατα... τα συζητάμε όλα αυτά και από την παρέμβασή σας κατάλαβα πως είστε ρεαλιστής πολιτικός, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί, διότι ακριβώς έχουμε μια συνθήκη και να θεώρηση μια συνθήκη ήταν τόσο δύσκολο να γίνει και γι' αυτό τα κρατημέλη αποφάσισαν να φτιάξουν μια νέα συνθήκη και όχι να αναθεωρήσουν την ισχύουσα. και ας ε, μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όσο γίνεται πιο σωστά αυτή τη νέα συνθήκη. Τώρα, αυτά που είπε η κυρία Σουόνσον από την ε, Σουηδία, συμφωνώ, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Ε, πώς μπορούμε δηλαδή να εμβαθύνουμε την εσωτερική αγορά, να καταργήσουμε τους φραγμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν και αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη για να μπορέσει να ε, ε, επιβιώσει η κοινή αγορά. Είναι όντως πρόβλημα εμπιστοσύνης. Χωρίς εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δεν θα έχουμε πρόοδο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα του υπερβολικού ελλείμματος. και του βιώσιμου χρέους, και όχι μόνο στην Ευρωζώνη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο από πολιτικές άποψεις και κάποιε φορέ είναι και πολύ οδυνηρό από κοινωνικές άποψει. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Εσωτερική αγορά. Η Κομισιόν το έχει προσπαθήσει πολύ. Το τελευταίο Συμβούλιο δεσμεύτηκαν οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων για να επιταχύνουν και να εφαρμόσουν νωρίτερα κάποια από τα μέτρα της ενιαίας αγοράς. Εάν δεν υπήρχε κομισιόν, να σας πω την αλήθεια, δεν θα υπήρχε και εσωτερική αγορά. Μπορώ να σας τα πω αυτά επί τη βάση της εμπειρίας μου 8 ετών σε αυτήν εδώ τη θέση. Πέρα από τις εθνικές μου εμπειρίες. Γιατί ο πειρασμό για τι κυβερνήσει είναι συνήθω να προσπαθήσουν να επιβάλλουν του δικού του κανόνε στου άλλου, αλλά να μην σέβονται του κανόνε οι ίδιοι πολύ κοινό πειρασμό. Υπάρχει μέγας κίνδυνος επανεθνικοποίησης των πολιτικών εάν δεν έχουμε κοινού θεσμού και κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε δει τόσες πολλές απόπειρε προστατευτισμού εντό τη Ένωση, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και πραγματική πίεση από όλε τις πλευρές και γι' αυτό χρειάζονται στεναρά όργανα στο κέντρο ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμο πεδίο και η εσωτερική αγορά που είναι το κόσμημα του θρόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αμφισβητείται. Ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαδικασία επιπαραβάση κατά του μεγαλύτερου κράτους μάλλον και κατά του μικρότερου, μάλιστα για το πολύ ευαίσθητο θέμα των υπηρεσιών, που ξεκίνησε διαδικασία για τη Γερμανία και την Ελλάδα. Ακριβώς την ίδια μέρα έγινε αυτό θα ήθελα να δω άλλους οργανισμούς που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο είδος αμεροληψίας και αντικειμενικότητας που ασκούν και η Κομισιόν στις ενεργές της και στις αξιολογήσεις της. Σε σχέση με την ερώτηση του κ. Σέρκας για την απασχόληση, νομίζω πως έχετε δίκιο βασικά. Συνήθως δίνεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις οικονομικές πτυχές και όχι στην απασχόληση. Και μπορώ να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. Το 2009 εγώ πρότεινα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να γίνει ένα συμβούλιο κορυφής για την απασχόληση. Δεν συμφώνησαν, δεν ήταν επίγον. Τότε ήταν η Περιτροπή Προεδρία, είχαμε η Τσεχική Προεδρία και είχαμε οργανώσει στην Πράγα με τον Πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας και τις προεδρίες πριν και μετά ήρθε ο Πρωθυπουργό της Σουηδίας και από την Ισπανία ήρθε ο Υπουργό Απασχόληση, ο κύριος Κορπάτσο, αν, θυμάμαι καλά το όνομά του. Δεν κατέστη τότε δυνατό γιατί δεν ήταν η σημασία, το σημαντικό θέμα η απασχόληση. Υπάρχει κάποια πρόοδος βέβαια για στο προηγούμενο άτυπο συμβούλιο παρουσίασα κάποιες πρωτοβουλίες για την απασχόληση για να κινητοποιήσουμε κονδύλια από το Κοινωνικό Ταμείο για τις 8 χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες με ταχύρυθμο ε, πρόγραμμα και έγινε μια πραγματική συζήτηση για την απασχόληση γιατί Θεωρούμε στην Επιτροπή ότι η απασχόληση θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά ως input στη γενική μακροοικονομική ανάλυση και συστάσεις. Σε σχέση με το Ευρώπη 2020 ήδη το ανέφερα. θα σας πω κάτι που είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και κυρίως για τους εθνικούς βουλευτές. Μόλις λάβαμε, ο Πρόεδρος Φανρόμπο και εγώ, για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μια επιστολή από 12 αρχηγούς κυβερνήσεων με κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη. Η επιστολή αυτή είναι πολύ βοηθητική, συμπεριλαμβάνει πολύ σημαντικές παρατηρήσεις, τις οποίες συμμερίζομαι. Αλλά ήταν ενδιαφέρον ότι ούτε μια φορά αυτοί οι αρχηγοί των κρατών δεν μίλησαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Δεν είναι παράξενο αυτό. Και αυτό έρχεται στο προηγούμενη παρατήρηση. Πλήρης αποσύνδεση μεταξύ της συζήτησης στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό σύστημα, α το πούμε, Βρυξέλλε, Στρασβούργο, Κομισιόν κτλ. και συζήτηση σε πολλά από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πιστεύω πως η δική σας δράση, η δράση των βουλευτών σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τόσο σημαντική. Διότι δεν μπορούμε να δούμε αποτελέσματα για μια στρατηγική που είπα και επαναλαμβάνω ομόφωνα εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα, όλα υιοθέτησαν εκείνη τη στρατηγική και στη συνέχεια όταν μιλάμε για εφαρμογή ή για επικοινωνία δεν γίνεται καμία προσπάθεια όσον αφορά την ιδιοποίηση αυτής της στρατηγικής που χρειάζεται τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και των εθνικών θεσμών πέρα από τους κοινωνικούς εταίρους της περισφαίρε, και άλλους σημαντικούς φορείς για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής. Πιστεύω πως είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη έγιναν κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεση του μηχανισμού προειδοποίησης. Αυτός βασίζεται σε ένα πίνακα επιδόσεων που ε, συζητήθηκε εκτεταμένα στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο. Είναι κάτι βέβαια το οποίο ετοιμάζεται σε επίπεδο επιτελείου. Είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση. Δεν είναι το α και το ω κάθε οικονομικής ανάλυσης, αλλά τώρα έχουμε ένα διαφανές εργαλείο στη διάθεσή μας για να κάνουμε μια ανάλυση. Κάποιοι ανέφεραν ε, την Γερμανία. Να σας πω ότι όντως Έχουμε ε, αναφέρει σε αυτή την ετήσια έκθεση ανάπτυξης ότι το 2012 θα γίνει οριζόντια ανάλυση και ε, ε, για τις επιπτώσεις των πολιτικών για τις μεγάλες αγορές και αυτό μπορεί να έχει σημασία για το γερμανικό πλαίσιο αλλά γενικά η Γερμανία ήταν μια πολύ, είναι μια πολύ επιτυχημένη περίπτωση πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει πετύχει η Γερμανία είναι ότι πριν από λίγο καιρό έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις που έδωσαν στη Γερμανία ε, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας, ώστε ολόκληρη η Ευρώπη να καταστεί πιο ανταγωνιστική σε σύγκριση με το τι συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου. για την Ελλάδα και το θέμα του κατά πόσο είναι δημοφιλής ή όχι οι μεταρρυθμίσεις. Συμφωνώ απολύτως. Πολύ δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα μπορεί μόνο να αντιμετωπιστεί μέσω αυξημένης ε, ε, ηγετικής ε, ικανότητας. Αυτό σημαίνει πως οι πολιτικοί σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πούν την αλήθεια και να θέσουν τον λαό ενώπιον των ευθυνών τους. Όλοι είστε και να δώσουν όμως και εναλλακτικέ. Εσείς είστε όλοι πολιτικοί. Ξέρετε ότι είναι εικόνα να υπάρχουν εναλλακτικέ. Ποια είναι η εναλλακτική. Εσείς πιστεύετε στην Ευρώπη με τόσο ψηλά επίπεδα χρέους η λύση είναι να γίνει ένα άλλο είδος φορολογικών, ε, δημοσιονομικών μάλλον κινήτρων για χώρες που είναι εξαιρετικά ευάλωτες που αυτή τη στιγμή είναι υπό τη στενή παρακολούθηση, την πολύ στενή παρακολούθηση των αγορών και των επενδυτών. Φυσικά και όχι. Γι' αυτό και χρειάζεται να προχωρήσει ο η δημοσιονομική εξυγίανση, η ευφυή δημοσιονομική εξυγίανση και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε στοιχεία για την ανάπτυξη. Και γι' αυτό τα όσα είπαν κάποιοι από εσά, τη σημασία δηλαδή τη σύνδεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού με του εθνικού, νομίζω ο κ. Σαλβατόρ Γκαρίγα το ανέφερε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε αρκετά μέσα αυτή τη στιγμή για να συμπληρώσουμε την προσπάθεια του εθνικού επίπεδου. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν χώρο πια δημοσιονομικό για να συνδυάσουν κάποια από αυτά τα μέτρα με κάποιες επενδύσεις. Και αυτό και σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις, ναι. Αλλά από πού θα έρθουν οι επενδύσεις, ειδού η απορία. Δεν έχουν περιθώριο πια οι χώρες είναι τόσο απλό το θέμα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τους κατάλληλους πόρους για επενδύσεις. Σας ανέφερα αυτό το ομόλογα έργων που σας συζητήσουμε στο Συμβούλιο. Είναι ένας τρόπος, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους να κινητοποιήσουμε επιπλέον κονδύλια που θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις στις υποδομές που να είναι κερδοφόρες μέσω και μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε με αυτές τις ιδέες. Κύριε Κίλαντ από την Πολωνία, σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας ε, και σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και ναι, η Πολωνία είναι πετυχημένη περίπτωση σε πολλούς τομείς τα όσα έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά λοιπόν κάθε ένα κράτος μέλος χωριστά και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που πολλοί ανέφεραν συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ισότητας των μεταρρυθμίσεων, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κάσα από το Ηνωμένο Βασίλειο έθεξε βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας. Θα είμαι ανοιχτό μαζί σας. Δέχεστε ή όχι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δημοκρατικό, δημοκρατικός θεσμός. Είναι σημαντική ερώτηση. Εγώ πιστεύω πως ναι, είναι δημοκρατικός θεσμός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες μας. Η Κομισιόν είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο. Εγώ έχω εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήμουν Πρωθυπουργός της χώρας μου πριν και πριν υπουργό και προηγουμένως βουλευτής εθνικός και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα δεν είναι και τόσο διαφορετικό γιατί στην ουσία μπορώ μάλιστα και να προχωρήσω. Δεν είναι δύσκολο να εκλεγεί κανείς, δεν είναι διαφορετικό μάλλον το να εκλεγεί πρωθυπουργό κανείς από ότι πρόεδρος της Επιτροπής. Όχι μόνο χρειάζεται να υπάρχει συνένεση όμω στο Συμβούλιο, αλλά μετά πρέπει να έχουμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μυστική ψηφοφορία. Βέβαια, άμα θεωρείτε ότι το κοινοβούλιο δεν είναι δημοκρατικό θεσμό, ε, τότε εντάξει. Έχει νόημα η παρατήρησή σα. Πιστεύω ωστόσο ότι η βάση τη δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο είναι το Κοινοβούλιο μα, όπω η Βουλή ε, των κοινοτήτων και βεβαίως ήταν ένα μεγάλο δώρο της βρετανική πολιτικής σκέψης και της βρετανική πολιτικής το δώρο τη αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και ζούμε στην Ευρώπη σε ένα σύστημα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δημοκρατιών μάλλον, όπου όλα τα κράτη-μέλη αντιπροσωπεύονται στο Συμβούλιο και οι πολίτες άμεσα εκλέγουν το Κοινοβούλιο. Και η Κομισιόν είναι υπόλογη, λογοδοτή στο Ευρωκοινοβούλιο. υπήρξε και η περίπτωση όπου η Κομισιόν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πρόταση μορφή. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία δεν έχει απόλυτα τα χαρακτηριστικά της εθνικής, αλλά είναι μια δημοκρατία, ε, δημοκρατία υπό εξέλιξη. Αν πιστεύουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να φτιάξουμε ένα σωστό σύστημα συντονισμού ανάμεσα στο εθνικό επίπεδο δημοκρατίας και το ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα αφήσουμε την πραγματική κυριαρχία όχι στα κράτη-μέλη, αλλά στις αγορές όπου οι οικονομικοί φορείς χωρί χωρίς ε, κανένα πρόβλημα θα επιβάλλουν το δικό τους, τους δικούς τους κανόνες. Στο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ακόμα και το πλουσιότερο κράτος μέλος μπορεί να συνεργαστεί επίσης όρις με την Κίνα ή με τη ΣΥΠΑ ε, Αν νομίζει λοιπόν κανένα κράτος μέλος ότι μπορεί μόνο του να το κάνει αυτό, ε, αυτοπατάται. Αν οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι θέλουν να μετράνε στον κόσμο, πρέπει να συμπληρώσουν την εθνική τους δημοκρατία με μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία και αυτό κάνουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Τα εθνικά μας κοινοβούλια, που όπως είπα στην αρχή, εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο για οποιοδήποτε προπολογισμό. Αλλά όταν ε, μοιραζόμαστε πληροφορίες με τα διάφορα κοινοβούλια, δίνουμε περισσότερη εξουσία, γιατί η ενημέρωση είναι εξουσία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος σε λύσεις που να είναι πολιτικά δημοκρατικές και που φυσικά θα έχουν και θετική ανταπόκριση. Αυτή είναι η βασική ε, ε, ε, ανησυχία όλων μας. Καθένας μας, άνδρας ή γυναίκα στην Ευρώπη, είναι η βάση κάθε δημοκρατικής νομιμότητας και αξιοπρέπεια, η αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους αγαπητούς συναδέλφους. Θα ήθελα κι εγώ συμπληρωματικά να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που έθεσε ο Πρόεδρος Μαρίνη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εκτός εθούσης όμως. Ναι, ναι, ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους μας. Α, βλέπω ότι έρχεται. Ε, κύριε Πρόεδρε ε, Μαρίνη, ε, αυτή τη στιγμή απαντώ στο πρώτο ερώτημά σας. Να συμπληρώσω την απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της συνεδρίασης για να εγγραφούν και να καταγραφούν αποφάσεις ή ληφθήσεις, για να υπάρξει ενημέρωση, είναι τεχνική σύσκεψη, είναι τεχνική συνεδρίαση. Η ιδέα είναι πολύ απλή και διαφανής. Θέλουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες ως προς την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, την κατάσταση των εθνικών οικονομιών, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πολιτικά μας εγχείρηματα και όπως το είπε άλλωστε και ο πρόεδρος Φαν Ρομπούι και πρόεδρος Μπαρόζο, θα έλεγα ότι πράγματι, όπως το υποδεικνύετε και εσείς ε, κύριε πρόεδρε Μαρίνη, στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε επί τη βάση κοινών σημείων αναφοράς. Είναι τόσο συνδεδεμένες οι οικονομίες ε, των χωρών μελών, ώστε όταν ε, καταρτίζουμε εθνικούς προϋπολογισμούς δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά, ε, την, ε, την αξία του ευρώ, την αξία που έχει το βαρέλι του πετρελαίου ή την, το, τις ισοτιμίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα αυτά είναι κοινά σε όλους μας και ίδια σε όλους μας. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη θεώρηση του συνόλου της Ευρώπης. Οι εθνικοί αντιπρόσωποι έχουν πλήρη δημοκρατική νομιμότητα ως προς τον εθνικό προϋπολογισμό και την εθνική οικονομική πολιτική. Χρειαζόμαστε να χρειάζεται να οργανώσουμε τη συζήτηση μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ ημών με ύψιλον και ε, ημών με ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε αυτή τη συνεδρίαση με μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Κοινοβουλίων και σήμερα το απόγευμα και μετά απόψε το βράδυ στο δείπνο και αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε με ανταλλαγές ε, μεταξύ ημών με ύψιλον. Γιατί? Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν τέτοιου είδους συναντήσεις είχαμε οργανώσει ήδη πριν από δύο χρόνια θα είχαμε αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά την ελληνική κρίση. Αν είχαμε την ευκαιρία να ε, ε, είχαμε κάνει έναν ειλικρινή, ανοιχτό, δημόσιο διάλογο με τους ε, ε, εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με τους εκπροσώπους των άλλων κοινοβουλίων, τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Αν είχαμε οργανώσει μια τέτοιου είδου ε, εξέλιξη των εργασιών μας, ίσως θα ήταν διαφορετικό το περιεχόμενο της συνθήκης αυτής για τους προϋπολογισμούς οι εθνικοί αντιπρόσωποι θα είχαν μπορέσει να εκφραστούν εκ των προτέρων, θα είχαν μπορέσει να συμβάλλουν στη βελτίωση της διατύπωσης της συνθήκης και έτσι θα, θα είχε ευκολυνθεί η κύρωση ε, της συνθήκης αυτής ε, σε όλες τις χώρες ε, μέλη οι οποίες προσχωρούν σε αυτή την συνθήκη. Κανείς βεβαίως δεν βρίσκεται εδώ για να εκπροσωπήσει την Γερμανία και να την υπερεσπιστεί. Οι Γερμανοί μας φίλοι δουλεύουν πολύ. Ε, δουλεύουν τη Δευτέρα και ψηφίζουν τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ψηφίζουν το πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα και δεν θα τους λέγαμε φυσικά να έρθουν εδώ σήμερα και να τους παρεμποδίσουμε και να μην είναι σε θέση να ψηφίσουν αυτό το πακέτο στήριξης. Ωστόσο, ε, εάν θέλουμε να συντονίσουμε τις οικονομικές μας πολιτικές πέρα και μετά από τη σημερινή κρίση προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την οικονομική μας μεγένθηση και την ανταγωνιστικότητά μας τότε όλοι πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες όχι μόνο σε επίπεδο προϋπολογισμού ή δημοσιονομικής ε, εξυγίανσης αλλά και σε επίπεδο π.χ. ενέργειας ή άλλων ε, θεμάτων ορισμένοι μπορούν να δυσκολέψουν ή αντιστοίχως να διευκολύνουν τη ζωή των υπολείπων. Και αυτό το στόχο έχουν αυτού του είδους οι συσκέψεις, να ε, διευκολύνουν τη ζωή όλων μας. 20 ζήτησαν το λόγο, δεν μπορούμε βεβαίως να το λόγουμε να τον δώσουμε σε όλους. Θα χωριστούμε τώρα σε δύο ε, εργαστήρια. Από τη μία πλευρά η υπέρμαχη της ε, δημοσιονομικής λιτότητας και από την άλλη η υπέρμαχη της οικονομικής μεγέθησης και της καταπολέμησης της ανεργίας. Ε, αστευόμενος βεβαίως τα λέω όλα αυτά. Έχετε το πρόγραμμα γραπτός. Θα έχουμε ε, τους επιτρόπους ε, και Χάν θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις. Η κυρία Μπόουλς θα προεδρεύσει. Ε, η κυρία Μπερές, όχι, η κυρία Μπόλτς, ε, και η κυρία Περβόνς Μπερές θα προεδρεύσει ε, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, δίνω στις συναδέλφους τον κατάλογο με όλους αυτούς οι οποίοι ζήτησαν το λόγο και οι οποίοι δεν μπόρεσαν να το πάρουν. Θα τους δοθεί ο λόγος κατά προτεραιότητα στο δεύτερο μέρος ε, της συνεδρίασής μας. Ε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος σε λίγο.